στο Seance and Direct από την ομάδα των Πρασίνων και το ΕΛΚ ε, έχουμε ε, τις προτάσεις για ορισμό για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και επιτροπές. Ε, αν δεν υπάρξουν ε, θα εγκριθούν. Ο πρόεδρος ε, της